Και ερχόμαστε στι επεξηγήσει ψήφου για τι εκθέσει που ψηφίσαμε το πρωί και είναι και πολλέ. Λοιπόν, θα τηρώ αυστηρά το λεπτό που έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Και μετά θα κλείνω το μικρόφωνο. Έκθεση Μπού Σούτιλ, ο κύριος Ρούντε πρώτος, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε, η αναθεώρηση του κανονισμού του Frontex ε, που επιτηρεί τα εξωτερικά μας σύνορα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα κοινά εξωτερικά σύνορα υφίστανται πιέσεις και στον κανονισμό ε, προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Ειδικά την Άνοιξη ήταν τεράστιες οι πιέσεις τα εξωτερικά μας σύνορα είναι κοινά. Γι' αυτό το λόγο, πριν από δύο χρόνια στη Δανία, το κόμμα μου στην προεκλογική εκστρατεία τονίσαμε ότι θα πρέπει όλες οι χώρες να συμμετέχουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο αυτών των συνόρων. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα γίνει με το νέο κανονισμό και όχι μόνο επειδή είναι σημαντικό, ε, να τηρούμε τις προεκλογικές μας υποσχέσεις, αλλά γιατί τα εξωτερικά σύνορα αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλώς πρακτικό, έχει και πάρα πολύ μεγάλη συμβολική λοιπόν σημασία. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ήτολα, για επεξήγηση ψήφου, απουσιάζει. Οπότε και θα περάσουμε στον κύριο Μποργέζη. Επίσης απουσιάζει. Ο κύριος Φιντάντσα. Παρευρίσκεται. Ο κύριος Μαστέλα. Έχετε το λόγο. ένα από τα προνόμια που υπάρχουν σε αυτόν τον κοινό χώρο ε, είναι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ε, άρει, να έχουμε καταργήσει τα σύνορα. Βεβαίω, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλά χάρη και κράτη και κατόπιν τούτου είναι ε, πηγόντως απαραίτητο να υπάρχει και μια συντονισμένη προσέγγιση. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν κοινέ διατάξει, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και καλύτερο συντονισμό των προσπαθειών, να υπάρχει και καλύτερη κατανομή των πόρων. Το βασικό στοιχείο που αφορά στην συνεργασία συνεργασία είναι να υπάρχει αλληλεγγύη κυρίως απέναντι σε εκείνα τα κράτη ε, που είναι όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν αυτά τα κράτη είναι εκείνα που δέχονται κυρίως τις μεταναστευτικές ροές. Τούτο ισχύει κυρίως για την Ιταλία. Ε, σε τελική ανάλυση μετά από πάρα πολλές διαπραγματεύσεις μπορέσαμε να επιτύχουμε θαυμάσια αποτελέσματα με την έκθεση αυτή που αφορούν στη Frontex. Ε, προβλέπονται περισσότερα κονδύλια και εργαλεία έτσι ώστε η Frontex να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω και το, ούτε τον κύριο Πίρκερ. Οπότε θα περάσουμε στην έκθεση μας η Πιτάλκο και πάλι ο κύριος Ρόντε, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας αυτή και πρόκειται για την πράσινη βίβλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, χρειάζονται ε, ε, πολύ προσοχή και θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια στις εταιρείες που αξιολογούν και βαθμολογούν τις χώρες θα πρέπει οι οικονομικοί ελεγκτές να είναι και ανεξάρτητοι αλλά να δίνουν και ποιοτικά στοιχεία, να διατηρηθεί η ποιότητα. Η κυρία Μαγκίνες παρακαλώ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το ρόλο των ελεγκτών. Η Ιρλανδία είχε μια δύσκολη εμπειρία και ο Φρανκ Ράιαν ε, αμφισβήτησε το ρόλο των οικονομικών ελεκτών που οδήγησε ε, στην ε, κατάρρευση των τραπεζών. Ε, σε μια υπηρεσία διαχείρισης των κονδυλίων γινόντουσαν τα εμβάσματα και μεταφορές. Και ποιος είχε τελικά την ευθύνη να επισημαίνει ε, τους ε, πολύ μεγάλους κινδύνους όπως είναι ο εξαιρετικό κίνδυνος που συσσωρεύτηκε σε κάποιες Ιρλανδικές τράπεζες την περίοδο 2004-2007. Και βέβαια ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά το ρόλο και το έργο των οικονομικών ελεγκτών. Θα χρειαστεί να αλλάξουμε τους κανόνες και ε, χτες είναι χάρη τον Επίτροπο Μπαρνιέ ε, για τις παρατηρήσεις του για το γεγονός ότι πολύ λίγες ελεγκτικές εταιρείες σωρεύουν πολύ μεγάλη εξουσία. κύριος Χάναν, για ένα λεπτό. Μα ο ε, ε, ε, ορισμός και μόνο της αφροσύνης και της τρέλας είναι να επαναλαμβάνει κανείς τα λάθη του. Και βλέπουμε τι γίνεται στο καρτούν της οικογένειας Σίμψον, όπου ο Όμηρος συνέχεια παθαίνει ηλεκτροπληξία γιατί μεταφέρει διάφορα ηλεκτρικά συσκευές. Εμείς είδαμε ότι έχουμε πρόβλημα με την ολοκλήρωση και κάνουμε ακόμα περισσότερη ολοκλήρωση. Πρόβλημα χρέους, άντε να το αυξήσουμε και το χρέος. Το θέμα αυτό ε, είναι ένα ζήτημα που είχαν τα κράτη στο εσωτερικό τους και τι κάνουμε, διονγκώσαμε το κράτος ε, και ε, το κάνουμε ευρωπαϊκό. Δηλαδή δίνουμε αντί για φάρμακο φαρμάκι στον ασθενή και βλέπουμε κάποιες δυσάρεστες ε, αυτο, αυταρχικές συμπεριφορές. Καλά. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά ανησυχώ αυτούς που βλέπω να μας κυβερνάνε. Mr. Kelly, Κύριος Κέλλη, για ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω το εξής ε, ο τίτλος αυτής της έκθεσης δίνει την εντύπωση ότι ίσως ε, έχει περάσει κρίση, ότι έχουν εξαχθεί τα μαθήματα. Δυστυχώς όμως αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε αν είμαστε στο μέσο ή στο τέλος της κρίσης. Και προφανώς όσο πιο γρήγορα τελειώσει η κρίση τόσο καλύτερα. Υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να εξάγουμε κυρίως ε, σε σχέση με τα ε, λογιστικά και τους λογιστικούς ελέγχους. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Μακίνες, ανέλησε σε το θέμα αυτό. Θέλω να πω ότι χαιρετίζω την ομιλία του Πολωνού Προέδρου. Χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες αισιόδοξε πρόπτικες ε, γιατί όπως είπε, το θέμα δεν είναι μόνο να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά να διασφαλίσουμε τη μόνιμη σταθερότητα. Ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά για να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα γίνουν, ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερότητα διάρκειας. Ε, για την επόμενη έκθεση το λόγο ο κύριος Ρόντο και πάλι. Έκθεση ε, Μπαρό. Er Πρόεδρε, πράγματι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν περισσότερη φτώχεια από τους άντρες. Έχουν χαμηλότερες συντάξεις, ε, διατρέχουν κίνδυνο να παραμείνουν άνεργες ε, παρότι ε, απολαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση και ζουν και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι και αυτοί είναι πραγματικοί. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το πώς θέλει να εμπλακεί σε όλη αυτή την κατάσταση, αυτό ομολογώ δεν το κατανοώ. Η απάντηση είναι ειδικά μέτρα για τις γυναίκες. Εγώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν στην αγορά εργασίας ε, ίσοι και δίκαιοι όροι έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, ε, να έχουν ίσες ευκαιρίες, ε, να μπορούν να απολαμβάνουν σύνταξη γιατί θεωρώ ότι πραγματικά αυτό το θέμα των ίσων ευκαιριών είναι καταλητική σημασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη γιατί καθορίζει τη θέση των γυναικών ε, που φτάνουν κυρίως ε, στην ηλικία της ε, συνταξιοδότησης. Βεβαίω το πράττει με έναν τρόπο που το θέμα δεν τίθεται για ευρεία συζήτηση. Χαιρετίζω το γεγονό ότι του χρόνου θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Χρονιά Αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενές γιατί το θέμα αυτό είναι πρόβλημα αλλά είναι πρόβλημα κυρίως για τις νέες γυναίκες και του νέου άντρε γιατί χρειαζόμαστε κάποιοι να μας φροντίζουν και αυτοί το πράττουν καθώς μεγαλώνουν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αν η έκθεση αυτή ε, θέσει στο προσκήνιο το θέμα, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό το καθήκον. Η κοινωνία χρειάζεται περισσότερε συζητήσει ε, για το τι δικαιούμεθα ε, και για το τι μπορεί να πληρώσει η κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμεί να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μα. Ε, αυτά που γίνονται με τη λιτότητα καθιστούν το θέμα πολύ δύσκολο, αλλά με αυτή την έκθεση τουλάχιστον κάνουμε μία αρχή. Χαίρομαι γιατί ασχολείται το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά με τις γυναίκες που είναι κοντά στη σύνταξη. Νομίζω ότι η γύρανση του πληθυσμού θα πρέπει να είναι ενεργός γύρανση διότι το προσδόκιμο ζωής είναι ακόμα μακρύτερο. Η σημερινή ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος των ε, γυναικών, διότι νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σχέσεις απασχόλησης και θέσεις απασχόλησης έτσι ώστε οι γυναίκες και πάνω από τα 50 να μπορούν να απασχολούνται. Σε σχέση με το συνταξιοδοτικό θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει μέτρα εποπτείας έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές ε, εισφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διότι πολλές φορές οι γυναίκες έπρεπε να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους. Η κυρία Χάρκιν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως ε, δείχνουν πολλά αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή το χάσμα μισθών κατά 17,5% με εξέπληξε αλλά μεταξύ 50 και 59 οι γυναίκες έχουν μισθό που ανέρχεται στο 67% του μισθού των ανδρών για, για το ηλικιακό αυτό φάσμα, το οποίο είναι και το δικό μου. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις για τις ε, συντάξεις τους και σημαίνει ότι κατά τη γύρανση θα πρέπει να ζήσουν μια κατάσταση φτώχειας. Επίσης, πολλές φορές οι γυναίκες διακόπτουν την σταδιοδρομία τους και δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι εκεί που οι γυναίκες πρέπει να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να ζήσουν σε κατάσταση φτώχειας σε μεγάλη ηλικία. Δεν, δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Ρόντα γιατί νομίζω ότι αν το πρόβλημα ήταν τόσο απλό δεν θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Έκθεση Μακάρθη. Κύριε Ρούντι, έχετε το λόγο. Υπάρχει το θέμα της ε, διαμεσολάβησης ε, και των περιφερειακών ε, διαφωνιών και βλέπουμε ότι έχει σημειωθεί επιτυχία σχετικά με το θέμα αυτό σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Είναι μια εναλλακτική λύση, όμως Πρέπει να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για τη διαμεσολάβηση και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τις σχετικές έρευνες για τη διαμεσολάβηση και να λάβει τα μέτρα εκείνα τα οποία θα επιτρέπουν την ορθότερη εφαρμογή ε, για τη διαμεσολάβηση. Έκθεση Reimers, ε, Κύριε Ντότζ, κύριε Πρόεδρε. Ε, με τη δική μου την εμπειρία στη Βόρειο Ιρλανδία η modulation μπορεί να αφαιρέσει χρήματα από τους ε, γεωργούς. Ε, έτσι λοιπόν ε, το είδαμε αυτό να ισχύει πρόσφατα στη δική μου την περιοχή στην Βόρεια Ολλανδία. Ανάλογα με το σχέδιο που εφαρμόζεται μερικοί αγρότες μπορούν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Και η αλλαγή αυτή πρέπει να πούμε δεν υπάρχει απαραίτητα. Οι άμεσες πληρωμές ε, είναι καθοριστική σημασίας για όλους τους γεωργούς ε, στην Βόρεια Ιρλανδία. Οι ε, πληρωμές αυτές θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύκολο, να μπορούν να αντικείμενο ευκολότερης διαχείρισης και να διατίθενται σε όλους τους αγρότες. Πρόεδρε, ξεκινήσαμε σήμερα την ψηφοφορία ανακαλώντας τις παροχημένες οδηγίες και διαρωτώ πόσο ευρία είναι, πόσο ευρύ είναι το πεδίο εφαρμογής αυτών των παροχημένων οδηγιών. Παραδείγματος χάρη στη Γεωργία, πράγματι εκεί υπάρχουν παροχημένες οδηγίες ή η κοινή ελευθερική πολιτική που βασίζεται στο μαρξιστικό αξίωμα ότι όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους πόρους, πλουταρικές πηγές Όλα αυτά ε, βέβαια ε, υπό την προπόθεση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 27 ε, διοικήσεις ε, οι οποίες ε, περιλαμβάνουν και πάρα πολλούς αναποτελεσματικούς αξιωματούχους. Δέστε λοιπόν πόσες αναχρονιστικές πολιτικές υπάρχουν ακόμα. Αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Ακόμα και η ότι το μεγάλο είναι και ωραίο. Τότε το να πιστεύει κανείς ότι όλοι ε, θα πρέπει να είναι ε, πιο πλούσιοι ας πούμε με την Ελβετία. Αυτό δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ξεπεραστεί από τις τεχνολογικές αλλαγές. Νομίζω ότι έκανα, ότι κάνατε ε, λάθος γιατί αντί να πείτε resource είπατε resort. Τι εννοείτε. Μπάση περιπτώσει. Ζαντό, έκθεση Ζαντό. Ο κύριος Σούστα. Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε πρωτοβουλία υπέρ της πραγματικής μας οικονομίας σε μία δυσχερή περίοδο κρίσης θα πρέπει να γίνει αποδεκτή πλήρως, διότι θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην παγκόσμια αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ζαντό και τους Σκιώδης, διότι μας έδωσαν μία έκθεση η οποία δημιουργεί διαφάνεια στις επενδύσεις, χωρίς να επιβαρύνει τις ΜΜΕ. Ελπίζουμε ότι στα πλαίσια αυτά και άλλες χώρες θα δεχτούν αυτή τη συμφωνία αρκετοί άλλοι εταίροι έτσι ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τους οικονομικούς φορείς και για να μην υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε ένα τομέα που αποτελεί το 10% του παγκόσμιου εμπορίου και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Αντωνιώτσι τα βιομηχανικά προγράμματα κατά το ίμιση στις υπονάπτυξη χώρες την χάνουν υποστήριξης από τη, τις ε, διάφορους, διάφορους οργανισμούς εξαγωγών έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε το περιβάλλον. Θα πρέπει να δούμε όμως τα ποσοστά αυτού του φαινομένου, δηλαδή ποιο είναι το μερίδιο αυτού του φαινομένου στην αγορά. Αυτή η κατάσταση δεν συνάδει με την πολιτική μας υπέρ του περιβάλλοντος. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα έπρεπε να κρίνουμε το εύρος αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε τους κινδύνους, αλλά χρειάζονται πολύ πιο σαφείς κανόνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε χρηματικά αυτά τα σχέδια για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, ο κύριος Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε αν μια εταιρεία λειτουργούσε με το μοντέλο του να πληρώνει τους καλύτερους πελάτες της. Ε, θα Δεν θα ήταν ε, ε, πολύ επιτυχημένη, όμως εμείς αυτή τη στιγμή με τις πιστώσεις εξαγωγών ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Ε, όμως τα πράγματα δεν λειτουργούν πολύ καλά έτσι. Μέσα, στα, μέσα της δεκαετίας του 1971 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 36% του ΑΕΠ, το 2020 θα φτάσει στο 15%. Τι θα κάναμε αν θέλαμε να μεγαλώσει η οικονομία μας. το στοιχείο έρχεται από τους ε, αριθμούς της Κόμισιον. Ο Γκούντερ ε, Φερχόγγεν μίλησε για το κόστος συμμόρφωσης με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι 6 δις το χρόνο. Έτσι λοιπόν τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς είναι 100 ε, ε, δισεκατομμύρια. Αυτά είναι με τα νούμερα της Κομισιόν. φαίνεται λοιπόν από αυτό ότι είναι πέντε φορές πιο ακριβή η ενιαία αγορά από ό,τι είναι τα ωφέλη της Πρόεδρε, οι χώρε ε, δεν έχουν εμπορικέ σχέσεις με άλλες χώρες, είναι οι εταιρείε που το κάνουν αυτό. Το καλύτερο λοιπόν είναι οι χώρε να βγουν από τη μέση. Ερχόμαστε στην έκθεση Κόφερ, ο κύριος Ρόντογκαν. Οι πρώτε ύλε ε, και κυρίω οι σπάνιε γεέ αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για τι οικονομίε μα. Η έλλειψη πρώτων υλών η ίδια αποτελεί μεγάλη πρόκληση αλλά υπάρχουν επίσης ε, κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται σε χώρες που δεν λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγάλες τάσεις σε προστατευτισμού και αυτό αποτελεί αίτιο ε, πολλών προβλημάτων. Ε, ξέρουμε ότι πολλές φορές πόλεμοι οφείλονται στα κοιτάσματα διαφόρων ορυκτών ε, χρειάζεται λοιπόν η εξωτερική υπηρεσία διμερό αλλά και πολυμερό να ασκήσει πίεση στις χώρε αυτές ώστε να υπάρχει διαφανής και ισότιμη πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Με αυτόν τον μηχανισμό θα πρέπει να λειτουργήσουν οι αγορές. Ο κύριος Δεάντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θεωρώ πως ε, το κλειδί για μια κατάλληλη προσέγγιση σε αυτό το θέμα συνδέεται όχι μόνο με εσωτερικό, εσωτερική παραγωγή, θα πρέπει αυτό να ενταχθεί στις εμπορικές πολιτικές όπως και στις αναπτυξιακές. Με άλλα λόγια, οι ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα στάνταρτα εργασιακά θα πρέπει να αποτελούν το μήμα αναπόσπαστο όλων των ε, συμφωνιών. Ε, οι πολιτικές καινοτομίες που είναι στραμμένες στο να αναπτυχθούν ε, διάφορες δεξιότητες μέσω μιας μεγάλης ε, ενός μεγάλου φάσματος μέτρων όπως η χρήση των πρώτων ελών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ή ο σεβασμός ε, των ε, συμφωνιών με τους προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται επίσης ειδική πολιτική για την ανάπτυξη πολιτικών καινοτομίας. Είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός και καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πολιτική αυτή αποτελεί βασικό κριτήριο για τη δημιουργία του ανταγωνισμού. Είναι μια πρόκληση η οποία απαιτεί μια συνεκτική μακροπρόθεσμη πολιτική και να υπάρχουν ε, και μέτρα ε, τα οποία να αφορούν στη διαχείριση και εξόριξη των υλικών. Ας δούμε το θέμα της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης. Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε και την διαφάνεια των συνθήκων ε, που υφίστανται για νέα ε, μεταλλεία. Ε, γιατί το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από την πρόσβαση σε όλα τα πρώτες ύλες. Πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε μια κοινοτόμο πολιτική η οποία θα διασφαλίζει ότι διαθέτουμε ασφάλεια των προμηθειών. και η πρόσβαση είναι σημαντική. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, ε, ψήφισα υπέρ ε, της έκθεσης Βουτκόφερ όχι μόνο γιατί πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά αν δεν την ψηφίσουμε θα έχουμε χάσει ε, ως προς την εφαρμογή των ε, ιδεών μας ε, και των στόχων μας και αυτό θα ήταν ένα μεγάλο έλλειμμα. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τους επόμενους μήνες όχι μόνο θα σκεφτεί πώς θα θέσει το θέμα στην Κομισιόν αλλά θα σκεφτεί και ως προς τον έλεγχο της εφαρμογής ε, να δει πώς ε, γίνονται τα πράγματα, πώς εφαρμόζονται από την Κομισιόν αλλά και πώς ελέγχεται αυτή η εφαρμογή. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει στο μέλλον να προσέξουμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο κύριος Αντωνιώτση. Πρόεδρε, δέχομαι θετικά την έκθεση Μπουτικόφερ χρειαζόμαστε μια σωστή βιομηχανική βάση για την ανάπτυξή μας και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν διαθέτουμε πρώτες ύλε. Η έλλειψη κοινή θέση έναντι της παγκόσμιας αγοράς μας φύγει ιδιαίτερα ως προς τις σχέσεις μας έφνη με την Κίνα, διότι δεν έχουμε μία συνεκτική πολιτική. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία κοινή θέση ως προς τις πρώτες ύλε και ελπίζω να δοθεί συνέχεια στην θέση μας αυτή και η ΕΕΔ να μπορέσει να ενισχύσει την κοινή μας αυτή θέση. Η κυρία Μουρκνάιτε. Πρόεδρε, συζητώντας τη στρατηγική μας για τις πρώτες ύλες και επειδή ακριβώς ε, θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα απόβλητα είναι η πρώτη, είναι μια πολύ χρήσιμη πρώτη ύλη. Πολλά κράτη-μέλη ε, ποντίζουν ή απορρίπτουν πολλά απόβλητα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς βασιζόμαστε σε μεταποιημένα αγαθά. Γι' αυτό θα πρέπει την ανακύκλωση να τη δούμε σαν, ένα πολύ, σαν μια πολύ μεγάλη πρόκληση και δυναμικό. Εάν μπορέσουμε έτσι να απορροφήσουμε τις πρώτες ύλε, θα μπορέσουμε να προβάλλουμε ευεργετήματα για τις οικονομίες μας. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χρήσιμη και σημαντική αυτή η έκθεση γιατί οι επιχειρήσει μα χρειάζονται πρώτε ύλε, αλλά θα πρέπει να προτείνουμε ότι από τα, μία από τι πρώτε ύλε κλειδιά που δεν έχει συζητηθεί είναι η γη. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα τη ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και με την ενέργεια και με τα θέματα κλίματο. Και από τα, μία από τι μεγαλύτερε ανησυχίε παγκοσμίω είναι το θέμα της ε, αρπαγής τη γη, όπου μεγάλες, ε, μεγάλοι όμιλοι αγοράζουν γη στον αναπτυσσόμενο κόσμο με αρνητικές επιπτώσεις για τον κόσμο που κατοικεί εκεί και που εξαρτάται από τη γη αυτή. Και το θέμα της ε, ε, διαθεσιμότητας γης και της χρήση της γης είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και κυρίω για τον αναπτυσσόμενο χώρο κόσμο και για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρώπης και είναι τμήμα του θέματος των πρώτων υλών γιατί η γη σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτή που έχει μέσα της, περιέχει μέσα της τις πρώτες και γι' αυτό και το θέμα του ελέγχου της γης θα είναι όλα ένα και μεγαλύτερη σημασία γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη γη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε σε μια παγκόσμια αγορά που χαρακτηρίζεται από ψηλή πτυτικότητα των τιμών και από όλα ένα μεγαλύτερη, μεγαλύτερη επίπτωση της οικονομίας στις αγορές, δεν μπορώ παρά να δεχτώ θετικά τη δημιουργία ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις πρώτες ύλες και τονίζω με ευχαρίστηση ότι μέσω της σημερινής ψηφοφορίας εντοπίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά τις πρώτες ύλε. και ταυτόχρονα επιφυλάσσεται μια μεγάλη, δίνεται μάλλον μια μεγάλη προσοχή στις δυσκολίες ανεφοδιασμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στα μέτρα που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό το ότι τονίζεται η υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητές, ρήτρε, συγκεκριμένες ρήτρες για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών ευθυνών των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καταψήφισα την εκθεσή για την στρατηγική των ε, πρώτων υλών, γιατί κατά βάση η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι ένας τρόπος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόσβαση στις πρώτες ύλες ε, με οποιοδήποτε κόστος, παρά τις καταστροφικές συνέπειες που οι διαδικασίες εξόρυξης έχουν στις, στους γηγενείς. Όσο ήμουν στο Καζακστάν, είδα τις επιπτώσεις της Αρσελών Μετάλ, μιας πολυεθνικής, η οποία ε, εκμεταλλεύεται ε, σε μεγάλο βαθμό τους εργαζόμενους της ε, και τον τοπικό πληθυσμό. Η διπλωματία λοιπόν αυτή της βιομηχανίας προσπαθεί να θέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπηρεσία της. Η συζήτηση έχει να κάνει λοιπόν με το ρόλο των μεγάλων επιχειρήσεων και την επιρροή του μέσα σε, αυτή την, αυτό το θεσμικό όργανο και υπάρχουν πολλοί βουλευτέ που ε, είναι πίσω από αυτή την έκθεση και εκπροσωπούν αυτά τα συμφέροντα. Αντί λοιπόν οι πρώτε ύλε να υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων ε, πολύ πλούσιων ε, πολυεθνικών, καλό θα ήταν να είναι πιο δημοκρατική η χρήση του και οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιούν για να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο όλων. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση, ο κύριος Μιλάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή, διότι είναι μία έκθεση η οποία προτείνει συγκεκριμένες ε, πολιτικές στον ευρωπαϊκό τομέα. Θα πρέπει να ορίσουμε την αλία σε αυτό τον τομέα και αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την Αδριατική όπου συνυπάρχουν διαφορετικές χώρες στον ίδιο χώρο, δηλαδή ενδοκινοτικές και εξοκινοτικές. Επίσης, θα πρέπει να θεωρήσουμε σημαντικό τη δημιουργία ε, της ε, αστυνόμευσης των παρακτίων. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία των παράκτιων περιοχών για τους αλληλείς και για τους καταναλωτές. Έκθεση Ford. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι έγινε με το Deep Blue Horizon και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστροφές στις υπεράκτιες δραστηριότητες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτιμήσουμε τις ευθύνες των κρατών μελών, διότι χρειάζεται συντονισμός και στη Βόρειο Θάλασσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεκταθούμε και σε άλλες ε, χώρες. Ε, όποιος μολύνει θα πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο και χρειαζόμαστε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες γι' αυτό. Η κυρία Μορκονάιτε. Νομίζω ότι τη στιγμή που υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη πετρελαϊκών προϊόντων γίνονται και οι κατάλληλες εξορίξεις ή γεωτρήσεις. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εξορεκτικές δραστηριότητες στις περάκτιες περιοχές είναι, ε, οι γεωτρήσεις αυτές είναι απόλυτα αναγκαίες, αλλά επειδή γίνονται σε υπεράκτιες περιοχές είναι και πιο επικίνδυνες. Αυτό μας ε, το έδειξε η καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού και η κρίση του Deep Blue Horizon. Χαίρομαι διότι η έκθεση έχει εντάξει και τις δικές μου τροπολογίες. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι η μόνηση δεν γνωρίζει η σύνορα. Γι' αυτό θα πρέπει να οριστούν οι ίδιες αρχές και για τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τις τρίτες χώρες για τις αρχές αποζημίωσης όταν πρόκειται για ε, περιοχές που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά και την εκμετάλλευση και με τη μεταφορά. Ο κύριος Πυρίλο. Να σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Μέσω της σημερινής ψηφοφορίας σίγουρα προχωρήσαμε προς μια βελτίωση της ασφάλειας και των ε, ελέγχων των ε, δραστηριοτήτων ανοιχτή θαλάσσης στον τομέα των ανθράκων έτσι ώστε να αποφευθούν ε, ατυχήματα όπως αυτό που συνέβη το 2011 στην πλατφόρμα ε, του κόλπου του Μεξικού που κόστισε τη ζωή 11 ανθρώπων ε, και είχε τεράστιες ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δέχομαι την πρόταση συντονισμού για κοινωνική προστασία αλλά και για τη δημιουργία υπερεθνικής δομής. Εύχομαι επίσης να υπάρξει αύξηση της συνεργασίας ανάμεσα στους ελεγκτικούς οργανισμούς ώστε να καθοριστούν κοινέ προδιαγραφές ανεξάρτητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ πως είναι θετική η δημιουργία ε, μιας ελεγκτικής αρχής στην Μεσόγειο για τις ε, δραστηριότητες ανοιχτής θάλασσας. Ο κύριος Σας ευχαριστώ. Όντως υπάρχει ανάγκη για κοινή δράση για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στις, στην ανοιχτή θάλασσα ακόμα και αν υπάρχει μια αρχή για τη Βόρεια Θάλασσα όπου έχουν υπάρξει διάφορα πολύ επικίνδυνα περιστατικά χρειάζεται ωστόσο να ληφθούν ε, στεναρά νομικά μέτρα για την ασφάλεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των ανθρώπινων ζωών. Αυτό σημαίνει την εξασφάλιση της συνεργασίας με τους γείτονές μας και, κυρίως ε, μιλώ για τους μεσογειακούς μας ε, ε, Γείτονε, αλλά και τη Ρωσία και τις ΕΠΑ. Πιστεύω πως κοινά διαφανή μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικά ωφέλη και μεγαλύτερη ασφάλεια ταυτόχρονα και γι' αυτό υποστηρίζω το ψήφισμα. Ευχαριστώ κύριο Μπαρτολότσι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταστροφή που χτύπησε τον κόλπο του Μεξικού πριν από ένα χρόνο όθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί για την νομοθεσία που σχετίζεται με τις ε, πλατφόρμες ε, Εξόριξη ανοιχτή Θάλασσα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεσή του θέλησε να εκφράσει τη θέση του για το θέμα εγκρίνοντας ένα κείμενο που απαιτεί δυνατότητες τεχνικές και οικονομικές από τους φορείς στον τομέα αυτό και στόχο έχει να θεσπιστούν υψηλά προδιαγραφές ασφάλειας έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας της δραστηριότητες ανοιχτής θάλασσα. Όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε διεθνή συντονισμό και σε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα συνδυάζει την αριστεία που υπάρχει στον τομέα, στον επίπεδο των διαδικασιών και, θα δημιουργήσει, και δεν θα δημιουργήσει επιπλέον δομές γραφειοκρατικές που μπορεί να απομακρύνουν από την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση συγκεκριμένα μετά από την μεγαλύτερη ευθύνη ε, των ίδιων των επιχειρήσεων απαιτεί μηχανισμούς επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων και αυξάνει το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και γι' αυτό θεωρώ θετικό το αποτέλεσμα στο οποίο φτάσαμε χάρη στην προσαρμογή αυτού του κειμένου για το οποίο έχουμε εκφράσει την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στην έκθεση για κουδάκι. Καταρχήν ο κύριος Μαστέλα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την δυνατότητα των γυναικών να μπορέσουν να δράσουν στο χώρο εργασίας και να βοηθήσουν με συγκεκριμένα ε, μέσα έτσι ώστε να έχουν μία ολοένα και υψηλότερη, μεγαλύτερη συμμετοχική πορεία στον εργασιακό χώρο. Υποστηρίξαμε την έκθεση αυτή διότι αναγνωρίζουμε της ΜΜΕ και γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, διότι οι εργαζόμενες γυναίκες έχουν να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κάθε εργοδότης είχε διαφορετική πορεία, ιδιαίτερα ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και στην ε, επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών. Ο κύριος Ρόντε. Είναι... δύσκολο να μην συμφωνήσει κανείς με τις ε, βασικές ιδέες σε αυτή την έκθεση. Λέμε ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι επικεφαλής επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν ε, και αυτές οι επιχειρηματίες με μεγάλες δεξιότητες. Ε, ε, το να συμφιλώσει κανείς την προσωπική με την επαγγελματική ζωή είναι δύσκολο και γι' αυτό θα πρέπει στο Κοινοβούλιο και στη Κομισιόν να βελτιώσουμε τις συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως γιατί μιλάμε συγκεκριμένα για τις γυναίκες ως επικεφαλής επιχειρήσεων. Γιατί θα πρέπει καταρχάς ε, να έχουμε ένα πλαίσιο με καλές συνθήκες για όλους που θέλουν να γίνουν επικεφαλής επιχειρήσεων, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες. Η κυρία Ντότζ. Έφυγε. Η κυρία Μαγκίνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε που με καλέσατε. Μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να πω ότι ενώ επικεντρωνόμαστε στο θέμα των γυναικών και των επιχειρήσεων, το βασικό πρόβλημα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι η διαθεσιμότητα των ε, εχεγγύων. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, ε, υπάρχει πρόβλημα Ε, με τις πιστώσεις εφόσον υπάρχει δυνατότητα να ζητηθούν περισσότερες πιστώσεις. Ε, το θέμα είναι ότι δεν αρνούνται να δοθούν αυτές ε, οι πιστώσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλη γραφειοκρασία η γραφειοκρατία όταν κανείς καταθέτει αίτηση για ένα δάνειο που τελικά δεν περνάει η αίτηση και δεν υπάρχει και επίσημη αναγνώριση της άρνησης αυτής. Δηλαδή η ίδια η διαδικασία μέσα ε, στις τράπεζες είναι που τελικά είναι συνώνυμη μιας ε, απόρριψης. Ε, και αυτό είναι πιο σημαντικό από το αν μπορεί κανείς, αν είναι άντρας ή γυναίκα, να γίνει επιχειρηματίας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χαρτίν. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για συστάσεις σε αυτή την έκθεση οι οποίες προωθούν τις γυναίκες όμως είναι επωφελείς και για τις γυναίκες και για την οικονομία μας. Γιατί ε, Υπάρχουν δύο βασικά θέματα που πρέπει να τονίσουμε. Είναι το θέμα της κοινωνική ασφάλειας στη χώρα μου και σε πολλές άλλες. Αν είσαι επιχειρηματίας και χάσει τη δουλειά σου, δεν έχεις κοινωνική ασφάλεια ούτε δικαιώματα τέτοια. Ε, και γι' αυτό δεν απορεί κανεί όταν οι γυναίκε ιδιαίτερα είναι επιφυλακτικέ στο να φτιάξουν μια δική του επιχείρηση. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα των κρατών μελών που πρέπει να το εξετάσουν επιμελώς. Επίσης υπάρχουν και τα προγράμματα μικροχρηματοδότησης που αναφέρονται στην έκθεση αυτά δίνουν μικροπιστώσεις ε, μέχρι και 25.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνήθως που δεν έχουν πρόσβαση από, στις τράπεζες. Ε, στην χώρα μου, στην Ιρλανδία, υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και θα καλούσα όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα καλούσα τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο παρόμοιο εργαλείο κύριος Μακέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας σχετικά με την με το χαιρετισμό των ε, προσώπων από τον Καναδά. Κοιτάμε λοιπόν τις ε, τράπεζες και τις εταιρείε ε, που εναπλάκησαν στην κρίση και βλέπουμε ότι ήταν λίγες οι γυναίκες ε, που ήταν επικεφαλής επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει κάποιος σωματικός ή ψυχολογικός λόγος για το αν θα πρέπει και οι γυναίκες να είναι επιχειρηματίες. Είναι ξεκάθαρο και έχει καταδεχθεί ότι πρέπει να δίνονται οι ευκαιρίες για να διασφαλίσουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. φυσικά αν οι ε, Lehman Brothers ήταν λίγο Women Sisters, ε, αν ήταν γυναίκες δηλαδή αντί για άντρες, ε, θα ήταν αλλιώς η κατάσταση. Θα... Έχουμε λοιπόν τους πόρους, ας αφήσουμε τις γυναίκες να συνεισφέρουν και αυτές με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επιχειρηματικότητα. Η κυρία Κλάς είναι η τελευταία μιλήτρια. Το μικρόφωνο όχι εξαιτία των γεγονότων, αλλά ε, γιατί πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ε, δυνατότητα να έχουν διοικητικά συμβούλια ή να έχουν τα κράτη ως μετόχους. Είναι δύσκολο οι γυναίκες... Υπάρχουν μάλλον κανονισμοί που λένε ότι πρέπει οι γυναίκε να συμμετέχουν σε τέτοια συμβούλια, αλλά πρέπει αυτά τα συμβούλια πρώτα να γίνουν. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι γυναίκες να έχουν ιδιαίτερη υποστήριξη για να μπορούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ε, και να συνεισφέρουν στην οικονομία. Ε, κάνουν μικρά μικρά βήματα στην αρχή και θα πρέπει να έχουν χρηματοδότηση γι' αυτό. Στην πράξη ε, αυτό το πρόβλημα υπάρχει όταν κανείς γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας, χρειάζεται κάποια κοινωνική ασφάλεια ε, για ασφάλιση γι' αυτό πρέπει κανείς να βοηθήσει τις γυναίκες ε, σιγά σιγά να μπουν σε αυτό το ε, παιχνίδι της κοινωνικής ασφάλειας, ασφάλισης και σιγά σιγά να γίνουν ανεξάρτητες. Ευχαριστώ. Να πω πριν κλείσουμε στους νέους που μόλις έφτασαν πάνω στα θεωρία ότι λυπάμαι αλλά η πρωινή συνεδρία σταμάτησε νωρίς ε, γιατί ε, είχαμε μια μεγάλη ψηφοφορία η οποία επανήλθε ε, στην Επιτροπή. Θα σταματήσουμε λοιπόν τώρα και λυπάμαι γι' αυτό γιατί ξέρω ότι ήρθατε από μακριά και είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και λυπάμαι που δεν θα δείτε τελικά τίποτα εδώ μέσα στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας τουλάχιστον. Ε, ε, Λύεται συνεδρίαση και συνεχίζουμε στις 3.